Mes chers collègues, Αγαπητοί συνάδελφοι, la séance est ouverte. Άρχεται η συνεδρίαση. Προηγουμένως όμως και πριν περάσουμε στην ημέρη σε διάταξη θα ήθελα να πω ότι όλοι έχουμε συνέστηση της νέας τραγωδίας που έλαβε χώρα χθες στη Μεσόγειο ανοιχτά της Λιβύης και σίγουρα 700 άνθρωποι έχασαν και πάλι τη ζωή τους, άνθρωποι που έρχονταν προς την Ευρώπη προσπαθώντας να ξεφύγουν από την αθλειότητα, να γλιτώσουν από τον πόλεμο και ως ένδειξη συμπόνιας ε, και συμπαράστασης στα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και προς όλους αυτούς τους λαούς, θα σας πρότεινα να κρατήσουμε ενός λεπτού nous ne pourrons nous en Δυστυχώς ε, φαίνεται ότι θα έχουμε μια αλληλουχία λεπτό, υγιής γιατί φαίνεται ότι και ένα νέο ναυάγιο έλαβε χώρα με νέα θύματα και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος ε, της μετανάστευσης και απαιτείται και από τις κυβερνήσεις μας αλλά και από σύσο την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάληψη σαφέστερων δεσμεύσεων φυσικά και με οικονομικό αντίκρισμα και δημοσιονομικό. Η κυρία Ματίας σας ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την αλληλουχία των λεπτών σύγκριση που μας ζητήσατε να κάνουμε να κρατήσουμε μετά από αυτές τις τραγωδίες που έλαβαν χώρα στη Μεσόγειο. Γιατί είναι η τρίτη φορά την εβδομάδα που πάνω από χιλιά άτομα έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα τη στιγμή που ξεκινούμε την ψηφοφορία, μη κυβερνητικέ οργανώσεις βρίσκονται έξω στην πλατεία του Λουξεμβούργου και ζήτησαν τη συνυποστήριξή μας και τη συμπαράστασή μας για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους αυτές τις εβδομάδες. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε έστω και για λίγο να βγούμε έξω στην πλατεία για ένα δεκάλεπτο σε ένδειξη συμπαράστασης προς όλα αυτά τα θύματα και μετά να περάσουμε στην ψηφοφορία. Νομίζω ότι δείξαμε την ελέγγυη μας κρατώντας αυτό το λεπτό σιγής. Όλοι έχουμε συνέστηση της εξαιρετικής σοβαρότητας της κατάστασης και νομίζω ότι ως Ευρωβουλευτές το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφράσουμε, να μεταφέρουμε και να δώσουμε σάρκα και οστά στις ανησυχίες μας και στη συμπαράστασή μας με την ψήφο μας και με την έγκριση πολύ πιο δαψιλών ε, οικονομικών μέτρων. Γιατί θα πρέπει να αφιερώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και να θέσουμε ως ύψη προτεραιότητα αυτό το θέμα της μετανάστευσης ε, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασιών. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν συμφωνείτε. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Καταρχήν τα πρακτικά της 26ης Μαρτίου είναι σωστά ή υπάρχουν αντιρρήσεις ή διορθώσεις. Δεν βλέπω παρατηρήσεις για τα πρακτικά, οπότε θα δώσω το λόγο στον Ρομπέρτο Γουαλτιέρη, γιατί εκείνος θα προεδρεύσει στις ψηφοφορίες. Γιατί όπως θα καταλάβατε, επιμερίσαμε έτσι το έργο, τα καθήκοντά μας, ώστε εγώ ανοίξω την έναρξη και το πέρα συνεδρίασης και το διάμεσο θα το αναλάβει ο Ρομπέρτο. Ευχαριστώ, Ζω. Μπορούμε να περάσουμε ευθύ αμέσω στην ψηφοφορία και να κάνουμε πρώτα απ' όλα έναν έλεγχο των μηχανημάτων. Δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ για τον έλεγχο των συσκευών. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν έχουν βάλει όλοι τις ε, κάρτες τους στη συσκευή. Κύριε Φερνάντες. Την περιμένω την, κάρτα μου. Θα φτάσει ε, ανα πάσα στιγμή. Okay. We can close. Τέλος ψηφοφορίας. Περνάμε λοιπόν στην κανονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία α. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία β. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία σ, γ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία δέλτα, D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Σίγματα F. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Θα ψηφίσουμε τρία ξεχωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας F. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 672. Ποιος είναι υπέρ. Γυρίστε στη σελίδα 14 του καταλόγου ψηφοφορίας παρακαλώ και τροπολογία 672. Θα έχουμε και μερικές μικροπροσθήκες. Για τελευταία στιγμή λάβαμε αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα. Παρακαλώ συγκεντρωθείτε. Τροπολογία 672 στη σελίδα 14. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 739 στη σελίδα 15 του καταλόγου ψηφοφορίας. Ποιος είναι υπέρ? Στην επόμενη σελίδα αυτή που ήταν προηγουμένως. Ποιος είναι υπέρ της 739? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία G. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία K. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 879, κοντ 39, ίδιες. Ποιος είναι υπέρ, τροπολογία 29, ε, σελίδα 29 του καταλόγου ψηφοφορίας παρακαλώ. Τροπολογίες 879, κοντ 39. Έχουμε διαφορετική αριθμή σελίδων. Καλά, δεν ξαναλέω σελίδες. Τροπολογία 879 και κοντ 39. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία L. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία M. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία N. Σε δύο τμήματα παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία O με προφορική τροπολογία από τους φιλελεύθερους ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ κατά ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία μόνο, όχι τη συμβαστική τροπολογία, μόνο την προφορική τροπολογία της Άλντε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική τροπολογία O, ο μικρόν χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ? Όχι, δεν είναι σε τμήματα. Ποιος είναι υπέρ της O, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 1019. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 1033 σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 1033. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε την τροπολογία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μια στιγμή, καταρχήν ανάψτε το μικρόφωνο. Για το 1033 δεν βλέπω δύο τμήματα εγώ στο κατάλογο ψηφοφορίας και τα έχω χάσει. Πού βρισκόμαστε. Ναι, τελευταία στιγμή υπευλήθη αυτό το αίτημα και μάλιστα τη δική σας πολιτική ομάδα, δεν κάνω λάθος, για να ψηφίσουμε σε δύο τμήματα, κάτι που έγινε. Ούτως ή άλλως και τα δύο τμήματα απορρίφθηκαν. Ξεκάθαρη διαφορά. Περνάμε στην τροπολογία 28 της Ρέτζη. 28 Ρέτζη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία π. Ποιος είναι υπέρ. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Q. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία R. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία S. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία τα φυπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ιού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, το είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία W. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Χ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Y. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Z. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία ΑΑ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΒ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AC. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AD ε, συμβαστική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AE. Υπέρ. ΑΕ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AG. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Ε, μάλλον πάμε κατευθείαν στο άρθρο 20, δεν έχουμε άλλες συμβαστικέ. Τροπολογία 1466, τροπολογία 1466, Αυτό μου λέει η γραμματή γιατί δεν υπάρχει συμβαστική πρόταση για το άρθρο 20. Θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε τις επιμέρους τροπολογίες για το άρθρο 20. 1466 τροπολογία. Αυτό μου λέει γραμματεία, δεν ξέρω αν διαφωνούν οι εισηγητές. Ε, αρνητικό πρόσημο έχει μπει. Όλες έχουν αρνητικό πρόσημο. Οπότε μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Όλες τις τροπολογίες για το άρθρο 20. Οι συγκεκριτές είναι κατά. Οπότε ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. AH, συμβαστική λύση, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AI, συμβαστική τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία AI α Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AJ. ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AK, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AL, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται AM ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία AN ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία AO ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία IP υπέρ, κατά, ποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία APBs, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε και συμβαστική τροπολογία APTER, ΑΠΒ δηλαδή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AP Quarter, δεν ξέρω πώς το προφέρετε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AQ. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AR. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AS. Ποιο είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ASBIS. Με προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε πρώτα την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε την ASB με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και να πάμε στο ASTER. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, κάπως ξαφνιάζομαι. Δεν ενημερώθηκε η ομάδα Άλντορ. Κάθε φορά που λέτε Μπίστερ και Κουάτορ δεν υπάρχει στην, στο κατάλογο ψηφοριών μας. Κάτι τέτοιο. Πρόεδρος. Αυτήν την ε, εκδοχή την μοιράσαμε στις τρεις. Και γιατί στις τρεις. Γιατί οι πολιτικές ομάδες ζήτησαν και λίγο μετά την προθεσμία να έχουμε κατατμήματα και ξεχωριστέ ψηφοφορίε, αλλά η μόνη αλλαγή που έχει γίνει είναι στα ονόματα των ε, ψηφίων. Όχι επί της ουσίας, δόθηκαν νέα ονόματα από τη γραμματεία. Πολύ λίγα. Μα κοιτάξτε, με συγχωρείτε πρόεδρε, αλλά ακόμη και αν ήταν μία μόνο ψηφοφορία, σε κοινοβούλιο είμαστε. Νομίζω ότι κάθε μέλος αυτού του σώματος πρέπει να καταλαβαίνει τι ψηφίζει δεν είναι απλώς θέμα ονοματοδοσίας. Ε, εδώ στο κατάλογο ψηφοφοριών μας δεν έχουμε καν τους ίδιους αριθμούς για την ψηφοφορία. Όπως επανέλαβα, εμείς μοιράσαμε αυτό το κατάλογο ψηφοφοριών σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Έχουν ακριβώς τον ίδιο κατάλογο όλες οι πολιτικές ομάδες. Πρέπει να το έχετε εκτυπώσει, ε, αν είχατε το προηγούμενο, και έχει μοιραστεί ως τις τρεις με αυτά τα γράμματα ο λόγος για τον οποίο ε, καθυστέρησε είναι γιατί η δική σας ομάδα και κάποια άλλη ζήτησαν ε, επιπλέον ξεχωριστές ψηφοφορίες. Οπότε γι' αυτό έγινε. Αλλιώς θα ήταν ο δικός σας ο κατάλογος. Το αίτημα προήλθε από τη δική σας ομάδα και από άλλες. Αλλά μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν οι πολιτικοί σας σύμβουλοι. Αυτό το κείμενο απεστάλλει. Όλοι το έχουν από τις τρεις. Πρόεδρε, όχι. Επιμένω. Πρώτα απ' όλα εμπιστεύω τους συνεργάτες μου, όλους, και ο λόγος για τον οποίο έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ και έχουν γίνει όλα άνω κάτω είναι γιατί τους συμβαστικές τις λάβαμε Κυριακή βράδυ. Την επόμενη φορά η ομάδα Άλντε θα ζητήσει αναβολή της πληροφορία. Πρόεδρο ευχαριστούμε. Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις σας και θα το μελετήσουμε, θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε. AS ε, Υπέρ. Πρόεδρε. Ναι. Πρόεδρε, μπορείτε τουλάχιστον να μας δίνετε το χρόνο να βρίσκουμε αυτές τις τροπολογίες. Απλώς δεν τις έχουμε μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Η κυρία Γκουλάρ έχει απόλυτο δίκιο. Συμβιβαστική AS e για το ε, εκτιμώντας 14 α. Δεν το έχουμε, δεν το έχουμε. Okay, I enough time. Σας έδωσα χρόνο. Υπέρ. Κατά. σες. Εγκρίνεται. Εάν χρειάζεται να τα διαβάζουμε. Συμβιβαστική. Μικρολάθος. Συμβιβαστική A, S, Κότερ για την αιτιολογική σκέψη 14C νέο. Να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εντάξει, να το διαβάσω, για να ελέγχετε. Πρόεδρε συμβαστική AES Quarter για το νέο τμήμα της ε, για την Ανατολική Σκέψη 14C, 247, 249 και 18 Ήτρε. Και η Ανατολική Σκέψη Νέο, το ΕΨΙ θα πρέπει να καλύπτει ε, και αξιόγραφα εγγυήσει ή χρέο, νέα προϊόντα, για τι ανάγκε των επιμέρου προγραμμάτων και αυτό το ευρύ φάσμα προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπει στο ΕΨΙ να ε, προσαρμόζεται στι ανάγκε τη αγορά και να ενθαρρύνει τι ιδιωτικέ επενδύσει τα σχετικά έργα. Δεν θα πρέπει να είναι υποκατάστατο για την χρηματοδότηση της ιδιωτική αγοράς ή για τους φόρους των ε, ε, τραπεζών σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, αλλά να ε, λειτουργεί καταλητικά για τις ιδιωτικές επενδύσεις και να καλύπτει τις ελλείψει της αγοράς, ώστε να υπάρχει σωστή χρήση του δημόσιου χρήματος ως μέσου για την οικονομική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να κάνω, έτσι κυκλοφόρησε στις τρει. Πριν από δύο ώρες. Πρόεδρε, παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν έχουμε γνώση αυτών των συμβιβαστικών. Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στην πληροφορία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά ποια είναι αυτή η στιγμή που αποστήλατε αυτές τις συμβιβαστικέ στους πολιτικούς συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Τι ώρα να σας εξηγήσω. Το ίδιο κείμενο κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο. Η μόνη αλλαγή που έχει γίνει είναι ότι έχουν χωριστεί σε τμήματα. Μπις, τέρ, κότερ κτλ. Δεν έχει αλλάξει ούτε μία λέξη. Να δώσω το λόγο και στον εισηγητή, τον κύριο Φερνάντε. Να σας πω απλώς ότι αυτές οι τροπολογίες είναι οι ίδιες που έχουν μοιραστεί την Κυριακή. Δεν είναι καινούργιες συμβιβαστικές είναι αυτά που κυκλοφόρησαν την Κυριακή. Δεν υπάρχει τίποτε το νέο. Κύριε Μπούλμαν. Συνάδελφοι, είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Και αυτό που είπε και ο, και ο Προεδρεύων. Η διαδικασία αυτή απαιτεί να συγκεντρωθούμε. Αλλά έχουν εργαστεί όλοι μας οι συνεργάτες από το Σαββατοκύριακο για να μπορέσουμε να έχουμε τη σωστή ε, το σωστό κατάλογο ψηφοφοριών. Την περασμένη εβδομάδα και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Πέμπτη είχαμε ενημερώσει όλους για τις συμβαστικές προτάσεις και γνωρίζουν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ε, το τι συμφωνήθηκε με κάθε σεβασμό ε, ενημερώσαμε τους πάντες. Ε, έχουμε λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις όλων. Ε, παρακαλώ δείξτε λίγη κατανόηση. Η προσπάθεια αυτή με την πίεση χρόνου που έχουμε έχει υποχρεώσει τους συνεργάτες μας να εργαστούν νυχθημερών τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ενσωματώσει όλες τις παρατηρήσεις, όχι μόνο των πολιτικών ομάδων, αλλά και των επιμέρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ίσως τις τελευταίες αυτές ώρες ναι, έγιναν αλλαγέ στον κατάλογο ψηφοφοριών, αλλά είναι τυπική αλλαγή. Ε, νέα ε, σειρά. Δεν υπάρχει αλλαγή επί τη ουσία, όπω σωστά είπε ο συνσηγητή μου Φερνάντε, για το περιεχόμενο. Οπότε, παρακαλώ, δείξτε κατανόηση. Α προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε και ευχαριστώ όλου για την κατανόηση που θα δείξουν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Ριάντα. Ευχαριστώ. Δεν θα σας καθυστερήσω, αλλά ούτε εμείς λάβαμε αυτή την πληροφορία. Είναι πολλές λοιπόν οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί δεν έχουν ενημερωθεί. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουμε να ψηφίσουμε στο δυνατόν γρηγορότερα, όμως πρέπει να δείξουμε σεβασμό και στο δημοκρατικό δικαίωμα όλων μας να γνωρίζουμε τι ψηφίζουμε. Οπότε, είτε θα ψηφίσουμε στι τροπολογίε που ήδη γνωρίζαμε και θα ψηφίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο τρόπο. Πρόεδρος, θα συνεχίσω να δίνω το λόγο στου συναδέλφου, αλλά σα επαναλαμβάνω, έχω εδώ το mail που απεστάλλει με ακριβώ αυτό το κατάλογο ψηφοφοριών. Μπορώ να σα διαβάσω τα ονόματα των παραληπτών. Ε, οι ομάδε σα ενημερώθηκαν. Το έλαβαν το mail με το κείμενο. Επαναλαμβάνω ότι το μόνο που έχει αλλάξει είναι απλώς στα τμήματα ότι οι τροπολογίες άλλαξαν όνομα επειδή προβλέφθηκε ένα ξεχωριστό τμήμα. Δεν υπάρχει αλλαγή περαιτέρω. Εάν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορώ να σας διαβάζω την κάθε τροπολογία, αλλά καλό θα ήταν να συνεχίσουμε την πληροφορία. Ο κύριος Τόρβαλτς. Η σύγχυση προκύπτει και γεγονό ότι όπως είπε και ο συναργότος Μπούλμαν, έχουμε νέα ονόματα για τις διάφορες ε, τροπολογίες που πρέπει να ψηφίσουμε. Με τα ονόματα αυτά ε, μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς ψηφίζουμε. Δεν είναι σωστή η διαδικασία έτσι. Δεν είναι επικριτικό το σχόλιο για τον κύριο Μπούλμαν ή τον κύριο Φερνάντες. Έχουν κάνει τεράστια δουλειά. Την εκτιμούμε, αλλά Μπράβο και στους ίδιους και στους συνεργάτες τους. Δεν βλέπουμε όμως τι ψηφίζουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Μπούλμαν και τον κύριο Φερνάντε. Αλλά εάν δεν ξέρουμε τι ψηφίζουμε, δεν, δεν ξέρουμε πού έχει γίνει η αλλαγή, είναι πολύ δύσκολο. Επιμένω. Μιλάμε για αλλαγή στα ονόματα, αλλαγή στα γράμματα και του αριθμού μόνο σε ένα πολύ μικρό αριθμό τροπολογιών. Πολύ, πολύ μικρό. Αυτοί, αυτές οι λίγες τροπολογίες έχουν αλλάξει όχι, όχι όνομα, αλλά έχετε λάβει τον κατάλογο ψηφοφοριών. Δεν ψηφίζουμε κάτι που δεν έχουν λάβει οι ομάδες επισήμως. Ισχύει για όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το βλέπω και ως πολιτική κίνηση. Μόνο από μερικές ομάδες προέρχονται αντιρρήσεις. Όλοι λάβαμε τα ίδια, την ίδια στιγμή. Δημοσίω κιόλα. Αν θέλετε να το συζητήσουμε άλλη ώρα περαιτέρω, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Μπορώ να πάω πιο αργά, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε. Το θέμα έχει ε, αποσαφινιστεί. Μπορείτε να επιμείνετε αν θέλετε, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί το θέμα δεν είναι αν έχει στάλει ένα mail Κυριακή βράδυ στι πολιτικέ ομάδε. Είναι θέμα του εάν οι βουλευτέ είχαν το χρόνο να διαβάσουν αυτά που έχουν αποσταλεί. Πολύ λίγο χρόνο για να ετοιμαστούμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Κύριε Λούκε, το, το πρόβλημα Δευτέρα απόγευμα είναι πολύ αργά εάν το στείλατε Κυριακή βράδυ. Είναι ντροπή έχετε εγκρίνει την ημερήσια διάταξη. Και όλες οι πολιτικές ομάδες επίσης την ενέκριναν. Ε, ε ζητήθηκε να δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση. Είχατε τη δυνατότητα οποιαδήποτε πολιτική ομάδα ήθελε να σηκώσει το χέρι της και να ζητήσει αναβολή της τροπολογίας, της ψηφοφορίας, συγγνώμη. Δεν είναι τώρα η στιγμή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο καθένας που θέλει να ε, επηρεάζει την έκβαση της ψηφοφορίας. Είναι διαδικαστικό. Είναι πολύ σαφές. Είχατε το χρόνο Έπρεπε να έχετε δράσει τότε. Δεν μπορούμε τώρα να βλοκάρουμε την πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση θα λέω την ανάλογη ονομασία της τροπολογίας, όπως για την προηγούμενη, για να έχετε το χρόνο. Άμα θέλετε να μπορείτε να τα διασταυρώσετε. Αλλά δεν θα χρειαστεί. Είναι πολύ λίγε περιπτώσει. Νομίζω ότι κάνουμε θέμα κάτι που είναι πολύ μικρή σημασία. Ψηφίζουμε πάλι. Ψηφίζουμε την AS Quest. για την αιτιολογική σκέψη 14 Δι νέο. Βασίζεται στην έμπλη 15. Εντάξει, υπέρ. Ψηφίζουμε. AS Quinques, ε, αιτιολογική σκέψη 14D νέο. Βασίζεται στην ε, τοποποίηση της έμπλη 15. Δείτε την γνωμοδότηση της ΕΜΠΛ και δείτε το ε, υπαριθμό 15 και θα το βρείτε. Δεκατέσσερα D. Είχατε τον κατάλογο. Τώρα πρέπει να το έχετε βρει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική AT. AT υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική AU. AU, με συγχωρείτε, ε, AU για την αιτιολογική σκέψη 16. Αιτιολογική σκέψη 16, υπέρ. 16, 16, 1, 6. AU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AU bis αιτιολογική σκέψη 16α υπέρ κατά αποχές να σας δίνω και την ανάλογη τροπολογία. AU bis βάσει της CALT 6 συμβιβαστική που βασίζεται στην ΚΑΛΤ 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική AV. Αιτιολογική σκέψη 17. AV. Αιτιολογική σκέψη 17. Με συγχωρείτε, αλλά αν θέλετε, ε, ελάτε εδώ. Εγώ προεδρεύω και διαβάζω ε, ποιο είναι η σωστή τροπολογία. AV, Ετοιμική σκέψη 17. Καλύπτει την τροπολογία, ε, τις τροπολογίες 331, 332, 333, αυκο 9, ΙΜΚΟ 9, ΙΤΡΕ, ΕΜΠΛ 23, ΙΤΡΕ 25. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. AW. Αιτιολογική σκέψη 18. Καλύπτει την 8, 349, 350, 351, 354, 355 ή 328. Αυτές είναι πληροφορίες που τις είχατε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 359 με προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε πρώτα την προφορική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σε αυτή την περίπτωση δεν με επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Πάμε στην συμβαστική AX. Η τηλεοκή σκέψη 19. Καλύπτει την 306, 8 και την έμπλη 25. AX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 382 382 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AY για την αιτιολογική σκέψη 20 Στηρίζεται στην τροπολογία 383 μόνο. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AYB για την αιτιολογική σκέψη 20α. Στηρίζεται στην τροπολογία 380, 381 και E332. Συμβαστική τροπολογία AYB. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται AYTER στη στην αιτιολογική σκέψη 20β καλύπτει τις τροπολογίες 385, 389, Τραν 11, άγρι 12 και Έμπλη 27. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές της AYTER, αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία AY Quarter για την αιτιολογική σκέψη 20C νέα. Ναι, Στηρίζεται στην τροπολογία 388 και καλύπτει και την τροπολογία 737. AY Quarter. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστικής τροπολογία, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AZ για την αιτιολογική σκέψη 21. καλύπτει τις τροπολογίες 9, 391, 394 ή 334. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία AZB για την αιτιολογική σκέψη 21α. Καλύπτει τις τροπολογίες Ρέγγι 11, 397, 38, Άμπλ 28. AZV, Β, ποιος είναι υπέρ, Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, Β, συμβαστική τροπολογία BA, ποιος είναι υπέρ, κατά. Η συμβαστική τροπολογία BA αφορά τη αιτιολογική σκέψη 22. Νομίζω ότι αφορούσε μόνο το προηγούμενο το αίτημα. Τέλος πάντων, η αιτιολογική σκέψη 22 ε, και η σχετική συμβαστική τροπολογία καλύπτει 405 και 406 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της ε, συμβαστικής τροπολογίας BA. Το σημαντικό είναι να βρείτε που βρίσκεται. Δεν χρειάζεται να ε, παραπέμπουμε πάντα στο προηγούμενο κατάλογο. Το θέμα είναι να βρείτε από ποιο αριθμό προέρχεται για να βρείτε γιατί τροπολογία πρόκειται. Δεν χρειάζεται να πείστε ότι πρέπει να αλλάξουμε το όνομα. Η κυρία Γκουλάρ, μία πρόταση κύριε Πρόεδρε. Μήπως θα μπορούσε ο κύριος Αρτουή να προεδρεύσει για να καθησυχάσουμε κάπως ε, τα πνεύματα γιατί φαίνεται ότι ε, αρνείστε το επιχείρημα μας ότι τα έχουμε χάσει λίγο, ότι έχουμε μπερδευτεί. Μα όχι, το λαμβάνω υπόψη και διαβάζω όλες τις τροπολογίες. Και αυτό που είπε ο συνάδελφος έδειξε ότι είχε βρει την, είχε εντοπίσει την τροπολογία. Στην προηγούμενη ψηφοφορία είχαμε διαφορετική αριθμίση. Γι' αυτό και τα εξήγησαμε όλα. Είναι σημαντικό τώρα όλοι να εντοπίζετε την ε, αντίστοιχη τροπολογία ώστε να μπορούμε να την ψηφίσουμε. Ψηφίσουμε λοιπόν τη συμβαστική τροπολογία BA. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται και περνάμε στην συμβαστική τροπολογία BB. Αφορά την αιτιολογική σκέψη 24 και καλύπτει τις τροπολογίες 420 και κοντ 8. 420 κοντ 8. Αιτιολογική σκέψη 24 και συμβαστική τροπολογία BB. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία BC για την αιτιολογική σκέψη 25. Καλύπτει τις τροπολογίες 10, 422, 423, 424, 427, 428, 431, κόντε 9, αύκο 15, ήτρε και Ρέγγι 13. Αιτιολογική σκέψη 25, συμβαστική τροπολογία BC. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 432 με προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την 432 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 38 της Ήτρε. Ή μάλλον συγγνώμη, στη συμβαστική τροπολογία BD. BD, συμβαστική τροπολογία, αφορά την αιτιολογική σκέψη, με ακούλπα λέει ο πρόεδρος, για την αιτιολογική σκέψη 26, καλύπτει τις τροπολογίες 11, 436, 438, 440, 442, 444, 449, κοντ 10, κουλτ 8, έμπλ 13. Συμβαστική τροπολογία BD για την αιτιολογική σκέψη 26. Ποιος είναι η τέρ. κατά, άποχες, εγκρίνεται. Ήτρε 38 τώρα, ψηφοφορία κατά θύματα ψηφίζουμε σε δύο τμήματα την τροπολογία 38 της ίτρε. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 38 Ήτρε, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία BE, αφορά την αιτιολογική σκέψη 27 και καλύπτει τις τροπολογίες 452, 453, 455, τραν 14 και ήτρε 39. Αιτιολογική σκέψη 27, επαναλαμβάνω συμβαστική τροπολογία BE. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Θέλετε να στη διαβάσω. Αιτιολογική σκέψη 27 δεν είναι καινούργια αυτή η αιτιολογική σκέψη από ό,τι ξέρω. Απλώς ε, τώρα τη λέμε συμβαστική τροπολογία BE. Άλλωστε δεν έχουμε άλλη τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 27. Είναι η μόνη συμβαστική τροπολογία για την 27. Εντάξει, να μην τη διαβάσω. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία BF για την αιτιολογική σκέψη 28 και στηρίζεται μόνο στην τροπολογία 12. Η συμβαστική τροπολογία BF ε, για το 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία BG κατά τμήματα. Αυτό ζήτησε η ομάδα μεταρρυθμιστών συντηρητικών. Στηρίζεται στην αιτιολογική σκέψη 29 η συμβαστική τροπολογία BG και καλύπτει τις τροπολογίες ε, 470, 71, 73, 475, 479, 481, 484, ήτρε 40, ΕΜΒΙ 21 και ΤΡΑ 15. Πρόκειται για την συμβαστική τροπολογία BG, αιτιολογική σκέψη 29, πρώτο τμήμα, Δηλαδή χωρίς τις λέξεις με ιδιαίτερη προσφυγή στο μέσο ευελιξίας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα της ίδιας συμβαστικής τροπολογίας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία BH, αφορά την αιτιολογική σκέψη 30 και καλύπτει τις τροπολογίες 491, 492 και κοντ 12. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία BI για την αιτιολογική σκέψη 31 καλύπτει της τροπολογίες 493, 495, 497, 98, 99, και 32 και κοντ 13. Συμβαστική τροπολογία BI. για είναι υπέρ, αιτιολογική σκέψη 31. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία BJ για την αιτιολογική σκέψη 32. 32 καλύπτει τις τροπολογίες 503, κοντ 14, κουλτ 10, ήτρε 9, ρέγγι 17, ήτρε 41. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία BK για την αιτιολογική σκέψη 33. Καλύπτει τις τροπολογίες 14, 506, ΕΜΒ 23 και ΚΟΝΤ 15. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία BL στην αιτιολογική σκέψη 34. Καλή τις τροπολογίες 517, ΚΟΝΤ 16 και ΤΡΑΝ 17. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία BM για την αιτιολογική σκέψη 35 στηρίζεται στις τροπολογίες, στην τροπολογία 523. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στα θεωρώντας, citations, Βρισκόμαστε στα θεωρώντας, εκτιμώντας. Τροπολογία 81, ποιος είναι υπέρ. Αφορά τον τίτλο. Πρώτα έχουμε τις αιτιολογικές αναφορές, το citation, και μετά θα πάμε στον τίτλο. θέλετε ψηφίζουμε και από κοινό τις αιτιολογικές αναφορές. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τώρα, 77 έχουμε πάει στον τίτλο. Τροπολογία 77. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 78 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 80, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση. Οπότε κηρύσω την έναρξη της ψηφοφορίας με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 66 υπέρ, 13 κατά και 9 αποχές. Αφήστε τα χειροκροτήματα για το τέλος. Έχουμε τώρα την ψηφοφορία νομοθετικού ψηφίσματος και πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος. 69 υπέρ, 13 κατά και 6 αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε την απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο με βάση τον, ε, το άρθρο 73. Ποιος είναι υπέρ. Και πάλι με ονομαστική κλίση πρέπει να ψηφίσουμε έτσι. Άρχεται ψηφοφορία ονομαστικά. Τέλος. 71 υπέρ, 6 κατά και 11 αποχές. Οπότε έχουμε συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, μπορούμε να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στους εισηγητές μας και να δώσω και πάλι το λόγο συμπρόεδρο, τον Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι άθλο επιτελέσαμε. Διότι η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της στις 13 Ιανουαρίου για την ε, προσαρμογή της νομοθεσίας και εμείς ψηφίσαμε το νέο κείμενο για να περάσουμε και σε με το Συμβούλιο. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τους, ε, τους μας, τον κύριο Μπούλμαν και τον κύριο Φερνάντες, το σύνολο των σχεδόν εισηγητών και όσες και όσους συνεισέφεραν στην ε, επεξεργασία του κειμένου αυτού. 3.000 τροπολογίες. Καταλαβαίνετε τι τεράστια πρόκληση ήταν αυτή. Τα καταφέραμε. Ήθελα να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για την ποιότητα των σχέσεων εμπιστοσύνη μεταξύ των επιτροπών μα, διότι κινητοποιήσαμε 13 επιτροπέ. Δύο μεικτέ, εικόν και ΒΑΤΣ, αλλά βάσει του άρθρου 54 του Αστρικού Κανονισμού ε, οι δύο είμαστε μέρες αρμόδιες και οι εννέα ε, βάσει του άρθρου 53. Ε, φέραμε εις πέρα στην πρόκληση αυτή και ήθελα λοιπόν να συγχαρώ θερμά και τους συνεργάτες μας από τη γραμματεία, εκτός από τους εισηγητές. Εξαιρετική η δουλειά τους και παρακαλώ τους χειροκροτήσετε. Δούλεψαν 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων και των Κυριακών. Δεν ήταν λοιπόν προφανώς απλό. Ο καθένας από εμά ήταν δύσκολο να έχει κατά νου την ε, λεπτομερή ε, έκφραση στο κείμενο. Ευχαριστώ τους εισηγητές, ευχαριστώ και τον ε, συμπρόεδρο Ρομπέρτο και μέσα σε μια ώρα πετύχαμε το στόχο μας πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Τώρα στις 24 Ιουνίου ελπίζουμε να έχουμε αίσιο πέρας ως τότε με τις διαπραγματεύσεις του συμβουλίου, και θα πρέπει ο καθένας μας να δείξει όλες του τις δυνατότητες της διαπραγματεύσευσης, ε, ε Πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα δείξει και αυτό την ίδια διάθεση συνεργασίας και ελπίζω να μην έχουμε μία συμπίεση των ε, ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων για να πετύχουμε τους στόχους μας του, ε, του Connecting Europe Facility και του Horizon 2020 αλλά να πετύχουμε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε συγκεκριτές θέλουν το λόγο. Ο κύριος Μπούλμαν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω και εγώ με τις ευχαριστίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συμφωνήσω και εγώ με τις ευχαριστίες και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον συνεισηγητή Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες σε ό,τι αφορά τις ευχαριστίες. Είμαστε από δύο διαφορετικές επιτροπές. Είχαμε και οι δύο την εντολή, όχι μόνο την εντολή των συναδέλφων από τις επιτροπές μας, αλλά και να λάβουμε υπόψη ε, την άποψη των πολλών ε, άλλων επιτροπών. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη και για τη συνεργασία. Να ευχαριστήσω τους Κιώδης και τους ε, υπόλοιπους συζητητές, όχι μόνο τον κάθε Λιναρμό των Επιτροπών, αλλά και, τον, ε, και τους συζητητές που μας έδωσαν γνωμοτοτήσεις. Έκανε εξαιρετική δουλειά και τελικά το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια των Επιτροπών των Πολιτικών Οικογενειών. Όπως σκοπεύαμε άλλωστε εξ αρχής. Να ευχαριστήσω επίσης τους πολλούς βοηθούς και να πω ότι συμφωνώ και με τον Πρόεδρο. δούλεψαν νύχτη ημερών, αλλά και τους μεταφραστές, όλους όσους ε, ασχοληθήκαν με το κείμενο αυτό. Εξαιρετική δουλειά. Και θα ήθελα να τονίσω εκ νέου ότι οι δύο γραμματείες, οι δύο γραμματείες που εκπροσωπούνται εδώ ε, δεν λυπήθηκαν ούτε τον παραμικρό κόπο για να μπορέσει να πετύχει αυτό το έργο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τέλος και τους δύο προέδρους που κατάφεραν να προεδρεύσουν σήμερα σε μια δύσκολη συνάντηση. Είναι ισχυρή εντολή, είναι ισχυρό το κοινοβούλιο και αυτή η ισχυρή εντολή θα μας βοηθήσει να φέρουμε σε έσω τέλος το έργο αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ. Και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου που βέβαια ήδη αναφέρθηκαν, αλλά για λόγους εξοικονόμησης χρόνου να συγχαρώ τον συνεισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν όλες οι εργασίες να ευχαριστήσω όλους τους και ε, εισηγητές για τη συνεργασία τους και να πω ότι είμαι βέβαιος ότι σε αυτήν την ε, έκθεση δεν αντικατοπτρίζουμε μόνο το πνεύμα και τη σκέψη του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά ε, αντικατοπτρίζουμε την άποψη της πλειοψηφίας. Γι' αυτό πετύχαμε συνένεση και ελπίζουμε να πετύχουμε και συνοχή. Ε, αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης, για μένα, μας ε, σημαίνει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διαπραγματεύσεις με αυτοπεποίθηση, με πυγμή. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί το πρόγραμμα Juncker το επιθυμεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Επαναλαμβάνω λοιπόν όσα ακούστηκαν προ προς τις ευχαριστίες και να πω ξανά ευχαριστώ, ευχαριστώ όσους συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια για τη σκληρή, τη δύσκολη δουλειά τους, κάποιες φορές με βίες ε, κόντρες, αλλά το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Γουαλχέρη, ευχαριστώ. Απλώ να θυμίσω ότι βάσει του άρθρου 73 η δημοκρατική ομάδα θα συναποτελείται από τον πρόεδρο, τον εισηγητή και του χιλιάδε εισηγητέ από τι καθήλυναμόδιε επιτροπέ και βάσει τη απόφαση τη διάσκεψη των πρόεδρων, η, βάσει του άρθρου 54 οι επιτροπέ Ήτρα και Τραν έχει γίνει λάθος εδώ, θα συμμετάσχουν στην δημοκρατική ομάδα όπως ορίζουν τα άρθρα 5B ε, και E και τα άρθρα 8, ε, 18 και βάσει του ε, άρθρου που ορίζει την ενισχυμένη αρμοδιότητα θα υποσυμμετέχει και η Επιτροπή Κουλτ με βάση των άρθρων 5, 4, α ως Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίσουμε τη λέξη της συνεδρίασης.